Il Presidente. Eccoci. Allora, la seduta è ripresa. Λοιπόν, συνεχίζεται η συνεδρίαση. Τα χθεσινά πρακτικά έχουν διανεμηθεί ήδη. Δεν ξέρω αν υπάρχουν παρατηρήσεις. Πρέγω. Νο. No?